το γεγονός ότι μείνατε μέχρι τέλους. Να ευχαριστήσω όλους όσοι έμειναν στην αίθουσα αυτή την ώρα. Να σας ενημερώσω ότι η επόμενη